ώστε να υπάρξει μια ευρύτερη δράση στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πίτροπε και όλους. Έχουμε 7 ψηφίσματα τα οποία έχουν κατατεθεί και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αμέσως μετά την επόμενη συζήτηση. Το επόμενο σημείο της ημέρας της διάταξης είναι το θέμα των διακρίσεων επί τη βάση καστών στις Ινδίες και ξεκινούμε με τους ε, εισηγητές της ε, πρότασης, κυρίως πρώτα τον κύριο Φαντάλεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δικαιολογημένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει μια συζήτηση σήμερα για την κατάσταση των λεγόμενων καστών στην Ινδία υπάρχουν 200 εκατομμύρια νταλίτ οι οποίοι βρίσκονται σε μια απαράδεκτη κατάσταση, εργάζονται κάτω από φρικτές συνθήκες και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για να μην σας χαλάσω το προϊόν, το μεσημεριανό σας. Και πολλές ε, από τις εκπροσώπους αυτού του πληθυσμού αναγκάζονται να εκδίδονται για να επιβιώσουν. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάνει προγράμματα, κάνει κανόνες, κάνει προσπάθειες υποτίθεται για να διορθωθεί η κατάσταση, αλλά αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι αυτοί οι οποίοι κατέστρεψαν τις κατοικίες των Νταλίτ, αυτοί που μετέτρεψαν τους Νταλίτ σε σκλάβους, αυτοί που εξώθησαν στην πορνεία τις γυναίκες Νταλίτ δεν διώκονται. Υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες ε, νταλίτ οι οποίοι βασανίζονται συστηματικά από την αστυνομία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εν πάση περιπτώσει ζουν χωρίς κανένα μα κανένα ανθρώπινο δικαίωμα και πρέπει κάτι να προσπαθήσουμε να κάνουμε για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Εμεί διαπραγματευόμεθα με την Ινδία για θέματα όπως το κλίμα, η ενέργεια, για θέματα εμπορικά και στα πλαίσια αυτών των συζητήσεων οφείλουμε να αναφερθούμε στην κατάσταση των Ταλίτ. Θα πρέπει να υπάρξει μια μεταρρύθμιση στην Ινδία έτσι ώστε η κατάστασή τους να μην χειροτερεύει συνεχώς. Πρέπει να τους προστατεύσουμε. Πρέπει να είναι προϋπόθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις σχέσεις της με την Τουρκία για τη σύναψη της νέας εμπορικής σχέσης. Με την Ινδία, συγγνώμη, για τη σύναψη της νέας εμπορικής σχέσης. Κύριε Γκέργια έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Το σύστημα των καστών υπάρχει σε πολλές χώρες της Ασίας. Ε, είναι θέμα συνδεδεμένο με την ιστορική τους παράδοση. Η διακριτική μεταχείριση και ο αποκλεισμός ε, κάποιων στρωμάτων του πληθυσμού είναι αποδεκτός κοινωνικά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι ανέγκυχτοι που ανήκουν στις ε, χαμηλότερες κάστες, ε, δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία και υπόκεινται σε εξευτελισμούς και καταναγκαστική εργασία. Μάλιστα Είχαμε μαζικό, μαζικούς βιασμούς και κακοποίηση παιδιών σε κοινότητες Νταλίτ. Βέβαια δεν έγινε επίσημη καταγραφή, καταγραφή τους, γιατί τα θύματα φοβούνται για τη ζωή τους και έτσι δεν καταγγέλουν αυτές τις παραβιάσεις. Και μάλιστα ε, το Σύνταγμα της Ινδίας προβλέπει ισότητα ευκαιριών ε, μεταξύ όλων των Ινδών. Υπάρχουν βέβαια στα ε, στα κείμενα αυτές οι διατάξεις, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται και εμπράκτως. Θα είναι δύσκολο να γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί δυστυχώς ε, το σύστημα των καστών είναι βαθιά ριζωμένο στην ε, ειδική παράδοση και ιδιαίτερα στις επαρχίες. Ελπίζω πάντως ότι και άλλες χώρες περιοχή θα διδαχθούν από το παράδειγμα της Ινδίας και θα αναλάβουν κάποιες νομοθετικές δραστηριότητες προκειμένου να πεταχθούν οι διακρίσεις εις βάρος κάποιων ε, κοινωνικών ομάδων. Για δύο λεπτά κυρία Λοχμπέντα. Ευχαριστώ. Οι Νταλίτ, αυτοί οι οποίοι ονομάζονται ανέγκυχτοι ή χωρίς κάστα, αποτελούν ένα τεράστιο τμήμα του πληθυσμού της ε, Ινδίας, περίπου 250 εκατομμύρια λόγω της κάστας μάλλον της έλλειψης κάστας τους, βρίσκονται κάτω από τεράστια πίεση και καταπίεση. Η Ινδία σε πολιτικό επίπεδο βέβαια έχει περάσει νόμους και έχει κάνει προσπάθειες για να δώσει ένα πέρας στην διάκριση επί τη βάση της κάστας. Αλλά βέβαια είναι πολύ περιορισμένη η, η επιτυχία της. Η απαξίωση των Ντάλιτς είναι κάτι το οποίο είναι εδρεωμένο στην παράδοση της Ινδίας. Με το ψήφισμά μας αναφέρουμε τον αριθμό των επιθέσεων που έχει γίνει, ιδίως πρόσφατα τον ε, Σεπτέμβριο στην Τάμπρα στο Χισάρ, όπου υπήρξε λαιλασία και εμπρισμός 268 σπιτιών σε κοινότητα ταντάλιτ χωρίς να υπάρξει καμία παρέμβαση της αστυνομίας. Η Ινδική κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό σε όλα τα επίπεδα να καταβάλουν προσπάθειες για να διατηρηθούν τα δικαιώματα των Ντάλιτ και ζητούμε να υπάρξουν οι απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες για να σταματήσει αυτή η διάκριση. Δυστυχώς, πολλοί Ντάλιτ έχουν αποδεχτεί αυτήν την περιφρόνηση εναντίον τους. Είναι έτοιμοι να δέχονται την ταπείνωση σαν να είναι η φυσιολογική τους μοίρα. Όχι όλοι όμως. Υπάρχουν αυτοί που αγωνίζονται από τους ίδιους του Ντάλιτ για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας μαζί τους και πρέπει να τονίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα υποστηρίξει αυτούς τους ακτιβιστές στη δράση της. Είναι τα θύματα αυτής της καταπίεσης και θα πρέπει να προστατευτούν από αυτούς που ασκούν αυτή την αποτροπιαστική βία και αυτή την σύγχρονη μορφή δουλείας εναντίον τους. Πρέπει να έχουν τις πλήρες να δίνουν τη πλήρη υποστήριξή μα. Ευχαριστώ, κύριε Λόχμπιλντερ. Ο κύριο Πρέδα, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το κείμενο του κοινού ψηφίσματος είναι συνέπεια πρόσφατων επεισοδίων που είχαμε στην επαρχία Ταμίλ Ναντού και στην επαρχία Χισάν. Τα γεγονότα αυτά έδειξαν τις τραγικές διαστάσεις των διακρίσεων εις βάρος ε, των Dalit. Η κυρία Λόχ Μπίλερ μας εξήγησε τι σημαίνει Dalit. Σημαίνει ανέγκυχτος. Ε, ανέγκυχτος είναι ο όρος που χρησιμοποιείται ε, συχνά όταν αναφέρεται κανείς στην ομάδα αυτή των Ινδών χωρίς κάστα. Και μάλιστα το θέμα πια έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις. Αναγνωρίζουμε με τις προσπάθειες της Ινδικής Κυβέρνησης για να καταργήσει τις διακρίσεις λόγω κάστας, αλλά θα θέλαμε να εφαρμοστεί και στην πράξη η νομοθεσία που υπάρχει στα χαρτιά και προβλέπει ισότητα. Βέβαια, η εξάλληψη των διακρίσεων είναι μια χρονοβόρα και μακροχρόνια διαδικασία, γιατί θα πρέπει να αλλάξουν η να αλλάξει η νοοτροπία. Αλλά πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν κάποια σημαντικά βήματα πρόοδου. Η Ινδία χρειάζεται και μια ανεξάρτητη αστυνομία, αδιάφθορους αστυνομικούς. Θα πρέπει οι αστυνομικοί να καταγράφουν τις καταγγελίες που γίνονται από θύματα τέτοιων διακρίσεων και να δίνεται συνέχεια. Και πιστεύω ότι και η Ειδική Βουλή θα μπορούσε να εγκρίνει ένα νομοσχέδιο για να εξελιχθούν οι εξευθυλιστικές μορφές εργασίας που πλήττει κυρίως αυτές τις ομάδες των ανέγκευτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Ακολουθεί η κυρία Σάγκε για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζεται η συστηματική απαξίωση και η δουλεία που αφορά εκατομμύρια Ινδών. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα σε σχέση με <clears throat> αυτά τα πρώτα μέτρα που έχουν πάρει οι Ινδικέ αρχές. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα. Ελπίζουμε ότι η νομοθεσία η οποία προτείνεται έχει υποβληθεί στο Ινδικό Κοινοβούλιο θα δώσει πράγματι προστασία στις πιο τροτές ομάδες του πληθυσμού. Πρέπει να εξασφαλιστεί και η ασφάλεια αυτών οι οποίοι καταγγέλουν διακρίσεις εναντίον τους και αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτές τις παραβιάσεις δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να έρθουν ενώπιον δικαστηρίων. Θα πρέπει να έχουμε υποστήριξη αυτών των ατόμων που είναι σε μειονεκτική θέση στην Ινδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τι προσπάθειέ τη ώστε σε τοπικό επίπεδο να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα και επίση θα πρέπει να προσπαθήσει να προσεγγίσει αυτέ τι μειονότητε, αλλά μέσα από ένα διεθνή διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ινδία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα τη διάκριση και των καταχρήσεων εναντίον των Ντάλιτ. Όλο ο κόσμο βλέπει με μεγάλο ενδιαφέρον την οικονομική ανάπτυξη τη Ινδία, αλλά συγχρόνω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η πρόοδο αυτή και η ανάπτυξη αυτή θα αντανακλάται και στη βελτίωση τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κυρία Σάκη. Ο κύριος Μέρφυ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το σύστημα αυτό με τις κάστες είναι ένα αντιδραστικό υπόλοιπο της ιστορίας το οποίο επιβάλλεται από τις κυρίαρχες τάξεις της Ινδίας χρησιμοποιήθηκε και από τους Βρετανούς απικιοκράτες και χρησιμοποιείται και από τους Ινδούς καπιταλιστές σήμερα. Οι νόμοι δυστυχώς είναι ένα πράγμα στην Ινδία και η πραγματικότητα είναι κάτι το διαφορετικό. Οι νόμοι για τη βία εις βάρος των Νταλή τα γνωρούνται. Η αποκομιδή απορριμμάτων με χειρονακτικό τρόπο εξακολουθεί να είναι μονοπόλιο ουσιαστικά για τους ανθρώπους αυτούς. Η αποκομιδή αυτή αποβλήτων. Νομιμοποιούνται ουσιαστικά συνθήκες στην Ινδία οι οποίες δεν αποτελούν παρά μια βαρβαρική εκμετάλλευση των εργαζομένων είναι μια απλή μορφή βίαιης εκμετάλλευσης φτηνού εργατικού ε, δυναμικού. Υπήρξαν επίσης κάποιες αντιδράσεις από γυναίκες που εργάζονται σε κάποιες περιοχές του Ναμίλ Ναντού και ε, ε, πλέκουν υφάσματα ή ετοιμάζουν ρούχα για μεγάλες γνωστές επιχειρήσεις της δύση. Ε, πολλές φορές οι γυναίκες αυτές καταλήγουν στην αυτοκτονία. Η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Η ανάπτυξη της συνδικής οικονομίας που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ωφελεί μόνο μία μειοψηφία της συνδικής κοινωνίας. Υπάρχουν συνεχείς νεοφιλελεύθερες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που πιέζουν εκατομμύρια Ινδών στον αποκλεισμό και στην απομόνωση και ωφελούν μόνο τα κέρδη των μεγάλων καταστημάτων λιανικής πώλησης της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάποιες περιθωριακές ομάδες όπως η Νταλίτ θίγονται ακόμα περισσότερο από τα μέτρα αυτά και γι' αυτό θα πρέπει οι Ινδοί να κινητοποιήσουν όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχουν έτσι ώστε να ανακληθούν αυτοί οι ε, νόμοι. Ευχαριστώ κύριε Μέρφια. Ακολουθούν οι ομιλητέ εξόμενων πολιτικών ομάδων. Κύριε Κόρχολα, για ένα λεπτό πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ντάλιτ είναι το χαμηλότερο στρώμα στην Ινδία και το σώμα του, το τμήμα του πληθυσμού που υφίσταται τη μεγαλύτερη καταπίεση. Τον τελικό, τα, τους τελευταίους ε, μήνες υπήρξαν πολλές αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν για να βελτιώσουν την ε, κατάσταση των τάλιτ έχουν βουλευτέ στο Κοινοβούλιο και υπάρχουν και κάποιε ποσοστώσει για την κατάρτιση και την επαγγελματική του απασχόληση. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να παραμένουν στο περιθώριο. Επί τη βάση των στατιστικών, οι Ντάλιτ είναι η μεγαλύτερη μειονότητα στην ε, Νότια Ασία η οποία υποχρεώνεται σε πορνεία για να ξεπληρώσει τα χρέη της. μόνο 25% ε, των γυναικών ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η νομοθεσία και θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των Ντάλιτς στις, ε, στα σχολεία. Η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει τι απαραίτητε ενέργειε για όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κόρχολα. Ακολουθεί κυρία Κρετσού για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη διαμαρτυρία μου για τις διακρίσεις λόγω κάστας. Και μάλιστα οι γυναίκες υπόκειται σε διπλή ε, διάκριση γιατί αφενός είναι γυναίκες και αφετέρου δεν, έχουν και καμία, δεν ανήκουν σε καμία κάστα. Υπόκειται σε κακοποίηση, διακριτική μεταχείριση, βιασμό, δεν έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, οι ειδικέ αρχέ θα πρέπει επιτέλου να λάβουν κάποια μέτρα. Γιατί ένα στου έξι Ινδού είναι ντάλι, δηλαδή αποκλείονται από το σύστημα των καστών. Θα πρέπει η Ινδία να εφαρμόσει και εμπράκτο το σύνταγμα που απαγορεύει τη διάκριση λόγω κάστας. Επίσης, η θέσπιση ενός συστήματος ποσοστώσεων στην απασχόληση τους βελτιώσει την κατάσταση. Μάλιστα, είπα ότι εκπρόσωπος θα πρέπει ε, να, αναθέσει, να, να επισημάνει αυτό το θέμα στις διμερείς συζητήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας. Ο Γιούλαντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό προσπαθεί να αντιμετωπίσει την, ε, τις διακρίσεις οι οποίες δυστυχώς είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες και επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπων στην Ινδία. Η Ινδική κυβέρνηση θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπαθίες της για να εξασφαλίσει ότι αυτές οι διακρίσεις θα περατωθούν αμέσως. Περίπου 200 εκατομμύρια ντάλιτ στην Ινδία εξακολουθούν να ζουν κάτω από αποτροπιαστικές συνθήκες. Είναι υποκείμενα βίας, βιασμών, μάλλον οι θύματα βίας, βιασμών και άλλων μορφών διαβασανιστήριων Σύμφωνα με μία έρευνα, η Ινδία είναι μία από τις πέντε πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο για να ζει κανείς αν είναι γυναίκα. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν ε, <clears throat> συλλεγεί δείχνουν ότι είναι φρικτή η κατάσταση και η Ευρωπαϊκή Κομισιόν θα πρέπει να πάρει αμέσως μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτέ τις διακρίσει. Ευχαριστώ. Κυρία για ένα λεπτό, Σλιέτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σύστημα των καστών είναι ένα παλιό καταπιεστικό σύστημα, τελείως παροχημένο για τον 21ο αιώνα. Οι Ντάλιτ και οι Αντιβάζοι υπόκεινται σε σοβαρές διακρίσεις. Όχι μόνο δεν ανήκουν σε καμία κάστα, αλλά δεν έχουν και κανένα δικαίωμα. Θεωρητικά απαγορεύεται τέτοια διακριτική μεταχείριση, αλλά δυστυχώς στην πράξη ισχύει και ιδιαίτερες βάρος των γυναικών θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε κάποιους όρους στις δικές μας κλωστιφαντορικές βιομηχανίες ώστε να μην συμβάλλουν στην καταπίεση αυτή και καταστολή των τάλιτ. Είμαι ο μόνος εδώ που ε, έχει χειρονακτικά ε, καθαρίσει τουαλέτα στο κοινοβούλιο. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που το κάνουν 10 ε, ώρες τη μέρα που καθαρίζουν τουαλέτες ε, σε δημόσιους χώρους, σε τρένα ή χειρονακτικά μαζεύουν απορρίμματα. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να τεθεί ένα τέρμα σε τέτοια διάκριση. Ευχαριστώ κύριε Πάσκα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ο αγώνας εναντίον των παραδόσεων είναι πάντα δύσκολο σε οποιαδήποτε κοινωνία, ιδίως όταν σε αυτές οι παραδόσεις το σύστημα των καστών στην Ινδία είναι πράγματι βαθιά εδρεωμένα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλο το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε σε συνεργασία με τις Ινδικές αρχές να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον αποκλεισμό των Dalit και να, και να σταματήσουμε την λειτουργία του συστήματος των καστών. Ιδίως οι γυναίκες οι οποίες ανήκουν στους Dalit ή στους αντιβάσει έχουν να αντιμετωπίσουν μια τεράστια μορφή διακρίσεως. Όλα αυτά δεν είναι αποδεκτά. Είναι υποχρεωμένες να κάνουν εργασίες οι οποίες να τηγινές βρώμικες είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίζουν την ε, περιφρόνηση των άλλων καστών. Έχουμε πολλές περιπτώσεις όπως η πρόσφατη αυτή που αφορούσε τους ε, βιασμούς στην Τάβρα μια 16 χρονη Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια έκκληση ώστε το ταχύτερο δυνατό να εφαρμοστεί η νομοθεσία για τις κάστες στην Ινδία, ώστε τα μέλη της κάστας των Ταλίτ να μην τυχάνουν χάνουν ταπεινώσεων και διακρίσεων. Η ευθύνη για την προστασία των πολιτών ανήκει πάντα στην Ινδία είναι η Ινδία η οποία πρέπει να πάρει τι απαραίτητε αποφάσει και θα πρέπει να κατευθύνουμε τι κριτικέ μα στην κυβέρνηση τη Ινδία. Γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στου άλλου ομιλητέ εξ πολιτικών ομάδων. Κύριο Κέλλη, ένα λεπτό πρώτα. Ευχαριστώ. Η Ινδία είναι μία από τις μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου και αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερα θετικό. Προχωράει όμως οικονομικά αλλά όχι κοινωνικά. Και αυτό βέβαια εν μέρει είναι κατανοητό γιατί δυστυχώς παλές συνήθειες είναι δύσκολο να ξεπεραστούν. Οι περισσότερες κοινωνίες έχουν κάποιες δίσκαμπτες μορφές ιεραρχίας και αυτό δυστυχώς αποτελεί ένα πρόβλημα. Εδώ απαιτείται πολλής χρόνος για να αλλάξουν οι αντιλήψεις και θα πρέπει όμως παρόλα αυτά το θέμα να αντιμετωπιστεί. Ε, ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σύντομα είναι η μεταρρύθμιση των αστυνομικών αρχών, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κυρία Κόρχολα αναφέρθηκε στο θέμα της, της εκπαίδευσης γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ταλίτ παραμένουν ε, αναλφάβητοι και επίσης να σταματήσει και η απαράδεκτη πρακτική της χειρονακτικής απόσυρσης αποβλήτων. Ευχαριστώ κύριε Σρέπο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολλές φορές εντάξει ψήφισμα για την κατάσταση των καστών στην Ινδία. Είναι αποτροπιαστική η κατάσταση των ανέγκυχτων, των ανθρώπων που δεν ανήκουν σε καμία κάστα. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση της θέσης τους ε, και γι' αυτό ε, φταίει η Ινδία κυρίως γιατί ε, μας φλόμωσε στις υποσχέσεις, αλλά δυστυχώς δεν ε, τηρεί τις υποχρεώσεις της. Και οι βιαιότητες ε, που διαπιστώσαμε το τελευταίο καιρό εις βάρος Dalit δείχνουν ε, πόσο ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί στην Ινδία. Είναι σαφές ότι οι κυρίαρχες κάστες οργανώνουν βίες επιθέσεις εις βάρος κοινοτήτων Ντάλιτ. Και δυστυχώς οι ειδικές αρχές δεν παίρνουν στα σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις που έχουν να τηρήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να σεβαστούν τα δικαιώματα των Τάλι. Ευχαριστώ κύριε Ρέπο. Ο κύριος Πόσελτ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα των Ντάλιτς είναι το τελευταίο θέμα που αντιμετωπίζουμε σήμερα το, ε, αυτό το έτος, το 2012. Δεν είναι ένα περιθωριακό θέμα. Όπως είπε η κυρία Λόχ Μπίλντερ, απαιτεί την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια μάσα, μάσα ανθρώπων που υφίσταται τεράστια βάσανα. Εγώ όταν ήμουνα νέος θυμόμουν ότι η Ινδία σήμαινε φτώχεια. Σήμερα η Ινδία σημαίνει μια δυνητική υπερδύναμη η οποία θα ξεπεράσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να ισχύει αυτό εν μέρη. Είναι μια τεχνολογική δύναμη η Ινδία αλλά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα της φτώχειας των Ντάλιτ. Το γεγονός ότι, υπάρχει, ότι γίνονται εκτρώσεις των ε, γυναικείων εμβραίων, ότι υπάρχει υπάρχει άσκηση βίας κατά τον Τάλιτ, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και στην εταιρική μας σχέση με την Ινδία θα πρέπει να τα αναφέρουμε. Θα πρέπει να ενδιαφερθούμε για το μέλλον, για τη μοίρα των Τάλιτ, γιατί αυτό είναι χαρακτηριστικό, είναι εμβληματικό τη μοίρα τη Ινδία και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ενεργητικά όλα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Πόσελ. Ερχόμαστε στην οφθαλμοσυλληπτική διαδικασία. Η κυρία Γκούρμα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η διάκριση λόγω κάστα στην Ινδία είναι μια εξοργιστική πραγματικότητα, συγκλονιστική παρά τις, ε, θε, τις νομοθετικές διατάξεις που υπάρχουν. Ο κοινωνικός αποκλεισμός ε, των γυναικών Ταλή είναι ανησυχητικός. Υπόκειται σε διάφορες μορφές βίας και εκμετάλλευσης οι γυναίκες αυτές ε, και ενδοοικογενειακή βία. Δυστυχώς η προστασία είναι ανεπαρκής μια και το κοινωνικό περιβάλλον καθιστά δύσκολη την καταγγελία τέτοιων κακοποίησεων. Οι γυναίκες που καταγγέλουν υφίστανται και, ε, και εξευτελισμό από αυτούς που ποτέ πρέπει να τους προστατεύσουν, όπως είναι οι αστυνομικέ και δικαστικές αρχές. Έχουμε συνθήκες εργασίας όπως είναι η χειρονακτική αποκομιδή απορριμμάτων ή απάνθρωπες συνθήκες απασχόλησης μοιάζουν με μορφές σύγχρονης δουλείας. Επίσης τα κλωστήρια που παρέχουν νήματα σε ε, δυτικές εταιρείε ε, απασχολούν κόσμο με από απάνθρωπες ηθίκες. Θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι μορφές εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκούρμαϊ. Έχει κλείσει τη διαδικασία Catch the Eye και μπορώ να δώσω το λόγο και πάλι στον Επίτροπο κύριο Τσόλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποιεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην Ινδία τον Νταλίτ που δεν ανήκουν στις γνωστές κάστες παρά την ισότητα όλων των πολιτών που προβλέπεται από το Σύνταγμα οι διακρίσεις παραμένουν η κυβέρνηση της Ινδίας έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς θετικών διακρίσεων βλέποντας ποσοστώσεις για τις κάστες αυτές και την πολιτική τους εκπροσώπηση. 84 βουλευτές στην κάτω βαλή του Κοινοβουλίου προορίζονται και 15% για την ανώτατη εκπαίδευση και 15% επίσης για τις θέσεις στη δημόσια διοίκηση παρά τις θετικές επιπτώσεις τις οποίες είχε η ρύθμιση αυτή δημιούργησε και στρεβλώσεις και υπήρξε μια κάποια ενίσχυση του συστήματος των καστών κάτι το οποίο δημιούργησε στο εσωτερικό αυτών των καστών προβλήματα με την δημιουργία υποποσοστώσεων. Πρόσφατα υπήρξαν κάποιες ρυθμίσεις όπως ο νόμος του 99 έτσι ώστε να αποφευχθούν ε, ενέργειες εις βάρος αυτών των μελών όπως ο νόμος του 99 που απαγορεύει ε, την χειρονακτική ε, αποκομιδή αποβλήτων, κάτι το οποίο όμως δεν εφαρμόζεται με ικανοποιητικό τρόπο. Στο δημοκρατικό τοπίο της Ινδίας κάποια πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στο κοινοβούλιο ή σε κάποιες επιπλέον πολιτείες φροντίζουν την προώθηση αυτών των καστών. Έτσι δημιουργούνται ε, διακρίσεις και αυτά είναι θέματα τα οποία γίνονται αντικείμενο συζήτησης στα πλαίσια του διαλόγου και τακτικά, ε, που τακτικά έχουμε με τους Ινδούς ομολόγους μας. Ένας τέτοιος διάλογος προβλέπεται στις αρχές του επομένου έτους πάρα πολλά σχέδια τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται από τις τοπικές αρχές και έχουν σαν άμεσο στόχο την βελτίωση των συνθήκων ζωής των λιγότερο ευνοημένων τμήματων του πληθυσμού με μια συγκεκριμένη θα έλεγα αφορμή την καταπολέμηση του αποκλεισμού όπως είπα και την κοινωνική δράση. Υπήρξαν αρκετά ισχυρές πιστώσεις για την δυνατότητα πρόσβαση στην δικαιοσύνη, για την καταπολέμηση της ένδυας. Εκεί δόθηκαν 433.000 εκατομμύρια, ε, ευρώ. Το σύστημα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι βαθύτατα βέβαια αγκυρωμένο στην συνείδηση των Ινδών. Από την ανεξαρτησία και μετά η Ινδία έχει κάνει σημαντικά βήματα για την πρόοδο, προς την πρόοδο. Αν και παραμένουν όμως αρκετές περιοχές ε, ε, σκοτεινές ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως στηρίζει τις δράσεις της ε, κυβέρνησης της Ινδίας η οποία κάνει προσπάθειες και έχει ξεκινήσει αρκετές τέτοιες προσπάθειες. Όπως είπατε και εσείς άλλωστε στο τελικό έγγραφο, στα πλαίσια των συζητήσεων της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών δεν υπάρχει άμεση αναφορά στο θέμα των καστών στο σύστημα αυτό. Παρ' όλα αυτά, εφόσον η συμφωνία αυτή γίνει αντικείμενο έξυπνη θα έλεγα διαπραγμάτευσης όπως τα επιθυμούσαμε, θα βοηθήσει την Ινδία και κατά συνέπεια θα βοηθήσει και τις λιγότερο ευνοημένες μερίδες του πληθυσμού. Ευχαριστώ τον Επίτροπο κύριο Τσόλες. Έχουμε 7 ψηφίσματα για, το... για τη λήξη τη συζήτηση. Έχει τελειώσει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αμέσως. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία για τα 7 ψηφίσματα που